Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Έχω λάβει από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών ορισμένες ε, αιτήσει για διορισμό σε κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Ο κατάλογος θα προσαρτηθεί στα πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης. Εφόσον δεν υπάρχει καμία αντίρρηση μέχρι το, την έγκριση των πρακτικών, αυτοί οι διορισμοί θα θεωρηθούν ως οριστικά αποφασισμένοι. Διακόπτω λοιπόν τη συνεδρίαση μέχρι τις 9.